σε κανένα σημαντικό ζήτημα. Οπότε, ερωτώ την Κομισιόν, εσάς, γιατί επιτρέπετε στο Πεκίνο να κινείτε έτσι, ενώ διεξάγει μια παγκόσμια εκστρατεία κατά της δημοκρατίας. Είχαν υποσχεθεί στο Χονγκ Κονγκ ένα δικό του σύστημα διακυβέρνησης και τώρα υπαναχωρούν. Εάν δεν μπορούμε να ευσυστούμε τη δημοκρατία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δεν μπορούμε απλά να εκδίδουμε ανακοινώσει συμπαράσταση στι δημοκρατικέ δυνάμει του Χονγκ Κονγκ. Πρέπει να μπορούμε να δράσουμε κιόλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να χαράξει την δική της στρατηγική. Δεν συμφωνώ με την ψυχοπολεμική ρητορία που βλέπουμε από την Ουάσιγκτον. Όμως, όπως είχε πει κάποτε η Μάργαρετ Θάτσερ, όταν κάποιο βρίσκεται στη μέση του δρόμου, τον χτυπάει η κίνηση, τα αυτοκίνητα και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, πού θέλετε να βρίσκεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα η κυρία Ιντόια Βιλανουέβα Ρουίθ για ένα λεπτό. Χθε μιλήσαμε στο το κοινοβούλιο για το θάνατο του George Floyd. Είναι σημαντικό να ακούσουμε ε, τι συνέβη η, η, την, η επίθεση που, έλαβε, που δέχτηκε η πράσινη ευρωβουλευτή, η ρατσιστική επίθεση. Μην ξεχνάμε και του νεκρού στη Μεσόγειο. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο δικό τη έδαφο για να μπορεί να ζητεί ε, ευθύνη για όλου του Τζορτ Φλόιντ του κόσμου. Ε, να ζητάει ευθύνε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εξωτερική πολιτική που βασίζεται στον αφοπλισμό, να βασίζεται στη διαμεσολάβηση, στο να μην υπάρχουν κυρώσει, την πολυμερή προσέγγιση, ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, κλιματική αλλαγή στο Χονγκ Κόνγκ. Προσπαθούμε απλώ να υπερασπιστούμε το δικαίωμα διαδήλωση, αλλά αυτό ισχύει και για το Εκουαδόρ, την Χιλή, ε, την Παλαιστίνη ε, και βεβαίως ε, δεν μπορούμε να μην στυλιτεύουμε τις παρεμβάσεις του Τραμπ ή της Βρετανικής κυβέρνησης. Χρειάζομαστε αμοιβαία συνεργασία έτσι ώστε να μπορούμε να φτάνουμε σε συμφωνίες αλλά να φαίνονται και οι διαφορές που υπάρχουν. Όπως παντού στον κόσμο ε, χρειάζομαστε κάτι περισσότερο από μια απλή συμφωνία ελευθέρων, ελεύθερου εμπορίου που δεν ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Πουτζντεμόν. Μια λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμε είπατε εκπρόσωπε. Ο στόχος της, του Χονγκ Κόνγκ εδώ, ο στόχος είναι η Κίνα να σεβαστεί το Χονγκ Κόνγκ. Τι σημαίνει αυτό. Να γίνει σεβαστή, σεβαστό το διεθνές δίκαιο και να γίνει σεβαστό το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Το να κάνουμε την Κίνα να σεβαστεί το Χονγκ ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε, όλες, σε όλη τη χώρα και να δώσουμε μια ελπίδα στους Ιουγούρους, παραδείγματος χάρη που αυτή τη στιγμή είναι θύματα ε, και θρησκευτικών αλλά και εθνικών ε, διώξεων. Εάν Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς αρκείται σε λόγια ε, και σε φωτογραφική διπλωματία ε, χωρίς ε, καλύπτοντας ουσιαστικά τον εμπορικό εταίρο που είναι η Κίνα ε, τελικά δεν θα φτάσουμε ποτέ στην, στην αρχή του μία χώρα, δύο συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείξει για άλλη μια φορά στην περίπτωση αυτή ότι έχει κάποιες αρχές αλλά έχει δύο διαφορετικά σταθμά. Ε, και εγώ δεν εμπιστεύομαι ιδιαίτερα αυτήν την διπλωματία που έχει δείξει ε, πόσο ευάλωτη είναι απέναντι στις κινέζικες ε, ε, πιέσεις. Ε, βεβαίως ευχαρίστως να με εκπλήξετε κύριε Μπορέλη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο Άντριους Κουμπίλιους για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπορέη, βεβαίως και καταδικάζουμε αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή οι κινέζικες αρχές κατά της δημοκρατίας ε, και και σε ό,τι αφορά τι διεθνεί τη βεβαίω ε, δεσμεύσει για το Χονγκ Κονγκ. Και βεβαίω είμαστε στο πλευρό του λαού του Χονγκ Κονγκ στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του για την αυτονομία του. Βεβαίω και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πιέσει το Πεκίνο την ερχόμενη εβδομάδα. Όμω υπάρχει και ένα παράδοξο εδώ στι δράσει ε, των κινέζικων αρχών. Προσπαθούν να καταστρέψουν τη δημοκρατία στο Χονγκ Κονγκ, κάτι που καταδεικνύει ότι φοβούνται αυτό το μικρό, τη μικρή νησίδα δημοκρατίας. Συνήθως οι αδύναμες αρχές είναι αυτές που φοβούνται. Και αυτό μου θυμίζει κατά κάποιο τρόπο το πώς κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση ακριβώς είχε, ήταν αδύναμη σε επίπεδο ε, της αρχής και φοβόταν τη δημοκρατία. Ε, οι Κινέζοι αξίζουν να, είναι, να, να ηγούνται παγκοσμίω, αλλά πρέπει να μάθουν να μην φοβούνται τη δημοκρατία και πρέπει βεβαίω να μάθουν από τι δημοκρατίε του Κόνγκ και τη Ταϊβάν. Ευχαριστώ πολύ και τώρα τον λόγο έχει ο Μικ Για ένα λεπτό παρακαλώ. Τον περσμένο Νοέμβριο ε, έχει αποφάσει το ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Ρωσία να, να υπερασπιστεί ε, τα, τα, τα τις αλλά δεν υποστηρίζει ουσιαστικά το Χονγκ Κόνγκ. Πρόκειται για μια καμπάνια κατά της Κίνας και υπάρχει μια κοινοφοβία ε, και βεβαίως ε, έχουν δοθεί εκατομμύρια ευρώ στους ε, σε αυτούς που υποκινούν αυτές τις ε, ε επιθέσεις της, ε, της διαδηλώσεις του Χονγκ Κόνγκ. Στις ΗΠΑ υπάρχει ρατσισμός, υπάρχει δουλεία, ε, υπάρχουν περισσότεροι μαύροι στις φυλακές της ΗΠΑ σήμερα από ό,τι υπήρχαν σκλάβοι στο παρελθόν. Ο, οπότε δεν πρέπει να μιλάμε για τις διαδηλώσεις του Χονγκ Κόνγκ. Πότε θα γίνει μια συζήτηση για την Ιεμένη, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορούμε ε, να είμαστε υποτελεί ε, σε μια παράνομη ουσιαστικά κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν σέβεται τον νόμο στι ΗΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό ο κύριος Τόνι Λόπεθ. Εστούρης White, παρακαλώ. Αναρωτιέμαι τι κάνουμε εδώ στο το κοινοβούλιο ε, τι είμαστε ο Νοστράδαμος, συζητάμε για ένα ζήτημα όπως το θέμα του Ισραήλ, ένα ζήτημα που ακόμα δεν έχει λάβει χώρα, δεν έχει προκύψει. Γιατί συζητάμε λοιπόν για το Ισραήλ, ειλικρινά και εδώ βεβαίως ε, προφανώς μα έχει καλέσει εδώ η άκρα αριστερά, οι κομμουνιστές, έτσι να το συζητήσουμε αυτό. Υπάρχουν πολλοί λογικοί άνθρωποι και στου πράσινου και στου σοσιαλιστέ που μπόρεσαν χθε να πάρουν ε, μια διαφορετική θέση, παραδείγματο χάρη στο θέμα τη Ευρωπαϊκή Συμφωνία με το Ισραήλ. Ε, να φανούμε λογικοί. Γιατί συζητάμε λοιπόν εδώ, επειδή υπάρχουν κάποια αιμονή. Κάποια συνάδελφο εδώ από του Ποδέμου, δεν ξέρω ποιοι είναι, που μίλησε για τη Χιλή. Η Χιλή εδώ και χρόνια δεν είναι δικτατορία. Το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Κούβα, εκεί έχουμε δικτατορίε. Καταλαβαίνω βέβαια στην αιμονή σα ε, με τη δημοκρατία του Ισραήλ. Αλλά αλλάξτε κάποια στιγμή κι εσεί το τραγούδι σα. Αλλάξτε ε, το ποιηματάκι σας ε, εδώ μιλάμε με την είπα το εκπρόσωπο. Μιλάμε για ένα ζήτημα ε, το οποίο δεν είναι για να συζητηθεί. Ας συζητήσουμε όταν συμβεί για την ενδεχόμενη ε, προσάρτηση. Δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για προεκλογικέ δηλώσεις των Ισραηλινών αξιωματούχων. Στο μέλλον μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κυρία Μαρία Αρένα, για ένα λεπτό, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι λίγο περδεμένη γιατί μόλις είδα τα αποτελέσματα της χτεσινής ψηφοφορίας για τη συμφωνία την αεροπορική με το Ισραήλ. Και αναρωτιέμαι είναι διατεθειμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακόμα να υποστηρίζει την ε, πολυμερή προσέγγιση. Βλέπετε υπάρχουν διάφορες ε, δικήσεις που ε, φαίνεται ότι καταπολεμούν την πολυμερή διάσταση. 437 δεν θέλησαν χτες την πολυμερή αυτή προσέγγιση. Οπότε η παρέμβασή μου δεν έχει να κάνει τόσο με αυτά που μας είπατε κύριε Μπορέλ, γιατί πιστεύω ότι θαραλέα ε, πήρατε αποφάσεις όσον αφορά την ε, σύγκρουση αυτή Ισραήλ-Παλαιστίνης. Αναρωτιέμαι όμως για μας, για τη δικιά μας τη δυνατότητα που έχουμε. Μήπως ε, έχουμε διπλό λόγο, δίπλα μέτρα και σταθμά με την Κίνα, το Ισραήλ από ό,τι φαίνεται τελικά δεν είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε κάτι το οποίο αποφασίζεται σε διεθνές ε, επίπεδο. Γι' αυτό και είμαι κάπως συγχυσμένη κύριε Μπορέλ. Ζητάω συγγνώμη, αλλά βλέπετε το θέμα όμως είναι δικό μας. Εμείς πρέπει να το λύσουμε εδώ στη συνέλευση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ναταλή Λουαζό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σήμερα εδώ θέλω να εκφράσω μια έντονη ανησυχία μου. Βάσει του συνασπισμού που έφερε στην κυβέρνηση στο Ισραήλ ε, η τελευταία εκλογική αναμέτρηση, τελικά γίνονται δηλώσεις και κάτι το οποίο είναι παράνομο, μια ενδεχόμενη προσάρτηση η οποία είναι κάτι παράνομο και το οποίο δηλητηριάζει τελικά το σχετισμό δυνάμεων. Εμείς εδώ στην Ευρώπη, παρά τα όσα μας διχάζουν, παρόλα αυτά υπάρχει μια βεβαιότητα που μας ενώνει και αυτή είναι ότι η βία δεν ε, δικαιούται τα πάντα συμφωνούμε, έχουμε την κοινή πεποίθηση ότι το κράτος δικαίου πρέπει πάντα να υπερισχύει και να μην υπερισχύει το δίκαιο του πιο δυνατού. Και αυτό το λέω με όλη τη φιλία που έχω απέναντι στο Ισραήλ, γιατί η φιλία ακριβώς επιβάλλει και κάποια καθήκοντα. Και το λέω γιατί θέλω να στηρίξω τη δημοκρατία στο Ισραήλ. Γιατί θέλω να το πω όπως το έκανε και η χώρα μου όταν είδε τις Ηνωμένε Πολιτείε το να ξεκινάνε για λάθος λόγους πόλεμο στο Ιράκ και που είχε τόσο αρνητικές συνέπειες στη συνέχεια. Ο ρόλος ενός φίλου λοιπόν δεν είναι να σιωπά, αντίθετα είναι να ξυπνάει αυτόν ο οποίος κινδυνεύει τελικά να καταστραφεί από τις πράξεις του. Εμείς εδώ στην Ευρώπη γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη παρά με τους εχθρούς μας. Εσείς στο Ισραήλ έχετε τη δύναμη με το μέρος σας. Εξυπηρετηθείτε από αυτήν ακριβώς τη δύναμη και χρησιμοποιήστε την για να πετύχετε την ειρήνη. Και μην ξεχνάτε αυτό που έλεγε ο Ισάκ Ραμπίν, ότι ένας δυνατός λαός μόνο μπορεί να καταλήξει σε ειρήνη με τους αντιπάλους του. Λοιπόν, ακριβώς επειδή έχετε αυτή τη δύναμη με το μέρο σας, να είσαστε και δίκαιοι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο, ο Ερνέστ Ουρτασούν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η προσάρτηση που έχει ανακοινώσει το Ισραήλ των Παλαιστινιακών εδάφων προφανώ και πρόκειται για κατάφορη παραβίαση ε, του διεθνού δικαίου. Πρέπει να τα πούμε τώρα, Ακριβώ πριν συμβούνε. Δεν πρέπει να περιμένουμε να συμβούν. Εσά μπορεί να μην σα ενδιαφέρει το να υποστηρίξετε το διεθνέ δίκαιο, αλλά οι περισσότεροι εδώ μέσα και οι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε θέλουν. Ε, υπερισχύει το διεθνέ δίκαιο. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό τα συζητάμε τώρα από πριν. Ε, ψηφίσαμε χτες, ναι, την αεροπορική συμφωνία με το Ισραήλ, αλλά διαφωνήσαμε γιατί γιατί ακριβώς θέλουμε να εκφραστούμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον όσο κάνει το Ισραήλ. Εδώ συζητάμε εδώ και καιρό ε, για το βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέμε ότι ενισχύεται τώρα που αποσύρεται από τη διεθνή σκηνή Ηνωμένες όμως υπάρχουν τεράστιες συνέπειες από μια τέτοια απόφαση στη Μέση Ανατολή του Ισραήλ. Έχουν γίνει ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Διπλωματία που λέει ότι αν υπάρξει μια τέτοια, ε, ένα τέτοιο βήμα θα απαντήσουμε σε αυτό. Και όντω θα πρέπει οι διπλωματικέ δυνάμει να φροντίσουν σε όλα τα επίπεδα να μην συμβεί αυτό, αλλά να ξέρει και το Ισραήλ ότι αν το κάνει αυτό το βήμα θα υπάρχουν συνέπειε και ότι θα ξαναδούμε τις σχέσεις μας με το Ισραήλ έτσι και συμβεί κάτι τέτοιο. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας λοιπόν και να στηρίξουμε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στα ε, ΝΟΙΕ ε, και παντού, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην υπάρξει ένα τέτοιο βήμα. Είναι ένα θέμα που και από το ΝΟΙΕ πρέπει να απαντηθεί έτσι και προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο Πάολο Μπόρκια. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα πρέπει να δούμε τα γεγονότα. Έχουμε εδώ πέρα μια νομοθετική πρόταση η οποία θα πρέπει να υπακούει κανονικά στους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Οπότε με βεβαίω από αυτά τα οποία ακούω, αλλά φαίνεται ότι στις Βρυξέλλες έχουμε ήδη ξεχάσει πώς λειτουργεί η δημοκρατία και βλέπουμε ότι προτείνονται διαδικασίες οι οποίες ε, αμφισβητούν το πώς λειτουργούν στο εσωτερικό τους τα κράτη. Θα πρέπει λοιπόν όσον αφορά την ε, Μέση Ανατολή να δούμε το Ισραήλ και την ε, Παλαιστινιακή Αρχή γιατί βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονομερής. Ε, η φιλοδοξία δε αυτών των μέσων είναι να ε, μπορούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία και το Ιράν να κάνουν ό,τι θέλουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι έχουμε μονομερή πειρά κατά του Ισραήλ. Επιπλέον, με βάση τα σχέδια τη νέα Ελληνική κυβέρνηση. Όμω η κατάσταση είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι την παρουσιάζουν οι συνάδελφοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για περιοχέ οι οποίε ανήκαν στην εντολή τη Παλαιστίνη, η οποία είχε προοριστεί για μια πατρίδα του εβραϊκού έθνους. Ε, επί σειρά ετών ανήκαν στην Ιορδανία και το 1960 σε έναν αμυντικό πόλεμο περιήλθαν στο Ισραήλ και εξακολουθούν να παραμένουν εκεί σήμερα. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν και μόνο καλό είναι να μην μιλάμε για προσάρτηση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου και να λέμε τέτοια μεγάλα λόγια. Και πάλι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει το λάθος να διαλέγει μονομερός τη μία πλευρά. Θα πρέπει λοιπόν να μην είμαστε μονομερείς. Ε, η σύγκρουση αυτή χρειάζεται μεσολαβητές, όχι άτομα τα οποία νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Μονού Πίνεδα για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Μπορέλ, στις αρχές Φλεβάρη μας είπατε ότι η προσάρτηση Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ δεν μπορούσε να περάσει χωρίς την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν ξεκινήσει η πανδημία ήμουν στην Παλαιστίνη ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να σας πω ότι παρά την αντίθεσή σας θα, ε, ε, αυτό το σχέδιο εφαρμόζεται βήμα-βήμα χωρίς να κάνουμε κάτι. Η τελευταία ανακοίνωση του Ισραήλ είναι πιο σοβαρή έως τώρα. Μιλάμε για την προστάτηση σημαντικού μέρους Τη δυτική όχθη, το 1 τρίτο μεταξύ των οποίων και ε, η ίδια η πλαγιά του Ιορδάνη μιλάμε λοιπόν για ένα σχέδιο ε, η λύση δηλαδή των δύο ε, κρατών που αυτή τη στιγμή ε, ψυχοραγεί. Ε, δεν ξέρουμε τελικά τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι δηλώσει είναι καταπληκτικέ. όμως δεν οδηγούν κάπου, δεν χρησιμεύουν σε κάτι. Θέλω να σα θέσω ένα ερώτημα και να θα ήθελα να μου απαντήσετε κύριε Μπορέλ. Τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναγνωρίσει το κράτο τη Παλαιστίνης. Γιατί δεν ακυρώνεται η συμφωνία σύνδεση εφαρμόζοντα το άρθρο 2 με το Ισραήλ. Και γιατί δεν παρεμποδίζουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μα επιβάλλεται ένα, γιατί δεν επιβάλλουμε ένα εμπάργκο όπλων ε, ε, στο Ισραήλ, γιατί δεν επιβάλλουμε ένα εμπάρκο προϊόντων που παράγονται στα κατεχόμενα. Ε, δεν μπορούμε να ακολουθούμε τον νόμο του ισχυρού. Πρέπει να ακολουθούμε τον νόμο της προστασίας του αδύναμου. Χρειαζόμαστε ειρήνη, αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η Εύην Ιμτσίρ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μπορέλ, οι συνάδελφοι του ΕΛΚ αναρωτιούνται τι κάνουμε εδώ σήμερα. <laughs> Αλλά το ΕΛΚ ε, δεν φαίνεται να κάνει τίποτα σχετικά με την ε, προσάρτηση των πεδαφών των Παλαιστινίων. Δεν κάνει τίποτα για να προλάβει κάτι τέτοιο. Αν αφήσουμε το Ισραήλ να προχωρήσει με το σχέδιο αυτό, θα είναι μια τεράστια οπισθοδρόμηση σε σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία. Η περίπτωση να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει ε, για δύο κράτη ε, είναι πλέον, θα γίνουν πλέον μηδαμινέ. Ε, υπονομεύει λοιπόν την όλη διαδικασία κάτι τέτοιο, αυξάνει την πόλωση και βεβαίως τη βία στην περιοχή. Η προσάρτηση αυτή θα αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και βεβαίως αντιβαίνει και το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται αυτό το σχέδιο του Τραμπ της τη ε, της του Ισραήλ ε, αποτελεί συνέχιση ουσιαστικά της επέκτασης ε, της, ε, της, του Ισραήλ. θα ήθελα να πω τελικά τι σκοπεύετε να κάνετε επακριβώς απέναντι στα σχέδια του Τραμπ αυτά ε, και πώς θα σεβαστούμε τελικά τα θεμελιώδη δικαιώματα και στις δικές μας περιοχές και παγκοσμίω. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο για να κλείσει αυτή η κοινή συζήτηση για τα τρία αυτά θέματα. Ε, επιπτώσεις της κρίσης του COVID, ε, Hong Kong και η ενδεχόμενη προστάτηση της δυτικής οχθής ε, από τους Ισραηλινούς. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον το εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο, τον κύριο Ζωζέ Μπορέλ. Παρακαλώ. Έχουμε χρόνο. Πέντε. Πέντε λεπτά. Πέντε. Πέντε λεπτά είναι αρκετός χρόνος για να απαντήσω σε 33 ερωτήσεις νομίζω. Όπως αντιλαμβάνεστε οι απαντήσεις μου ε, δεν θα είναι επαρκής ε, όσο θα ήθελα. Πασεπτός χαίρομαι που συμμετέχω στη συζήτηση αυτή και καλό θα ήταν να, έχω και να έχουμε και την ευκαιρία ε, να υπάρχει μια περισσότερη διάδραση μετά τις απαντήσεις μου αλλά εν πάση περιπτώσει στο μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσω να απαντήσω τώρα για το Ισραήλ και την προσάρτηση ακούστηκαν πολλές και διάφορες απόψεις εγώ αυτό μπορώ να σας πω ε, κάποιος είπε ότι είναι αμφισβητήσιμο το κατά πόσο συνάδει με το διεθνές δίκαιο τι να σας πω υπάρχουν 25 από τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης που θεωρούν ότι εδώ υπάρχουν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μπορεί να κάνουν όλοι λάθος, αλλά αυτό πιστεύουν. 25 από τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης υποστηρίζουν μια δήλωση που αναφέρει ότι εδώ έχουν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Γιατί μιλάμε γι' αυτό τώρα. Μιλάμε γι' αυτό διότι δεν θέλουμε να συμβεί. Ε, δεν ξέρουμε ποια είναι τα σχέδια του κράτους του Ισραήλ. Δεν είναι έτσι τα γνωρίζουμε. Είναι δημόσια. Αποτελούν μέρος της ε, συμφωνίας της κυβέρνησης συνασπισμού. Μου το λένε εμένα απευθείας υπουργοί αυτής της κυβέρνησης. Το είπαν στον Γερμανό υπουργό που πήγε στο Ισραήλ. Ότι το ξέρουμε λοιπόν, το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε εδώ πολιτική στρουθοκάμιλου. Τι κάνουμε λοιπόν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε διπλωματικό επίπεδο να μην συμβεί αυτό το πράγμα να μην βρεθούμε προ αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει το κράτο τη Παλαιστίνη. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει κανέναν. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν κράτη, άλλα κράτη. Και το κάθε κράτο ε, κάνει τι επιλογέ του. Τι μέτρα θα πάρουμε. Α μην προδικάσουμε τι θα συμβεί εδώ. Α περιμένουμε. Βεβαίω ε, η θέση, η πλειοψηφία, εν των κρατών μελών και όχι η ομοφωνία Δυστυχώ ε, ε, δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει ομοφωνία διότι δεν υπάρχει είναι ότι εδώ υπάρχει παραβίαση του διεθνού δικαίου και προφανώ θα υπάρξουν επιπτώσει. Εμεί θέλουμε να αποφύγουμε να συμβεί αυτή τη στιγμή τώρα για το Χονκό και την Κίνα δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας ε, είναι αναγκαίο να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να γίνουν σεβαστές οι διεθνεί συμφωνίε ε, μεταξύ της Κίνας και ε, με, με της Κίνας και στα πλαίσια της συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο όταν έπαψε το Χονγκ να του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχει λοιπόν μια έντονη δραστηριότητα έτσι ώστε να πιστούν οι Κινέζοι να σεβαστούν τι δεσμεύσει του. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Κίνα, τα οποία θα μα απασχολήσουν στην ε, μελλοντική ε, Σύνοδο Κορυφή. Αναφερθήκατε σε πολλά από αυτά. Α επικεντρωθούμε σε ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο αναφέρατε πολλοί από εσά. Η κρίση έφερε μαζί της, το είπε και ο κ. Μπουτικόφερ, το είπαν και άλλοι, ε, ε, μας έδειξε την κρίση της αμερικανικής ηγεσία. Φάνηκε δηλαδή πως δεν μπορούσε να ηγηθεί ε, να ηγηθούν οι πολιτείες ε, της μάχης κατά της πανδημίας και βεβαίως υπάρχει μια αποδυνάμωση των διεθνών οργανισμών. Έτσι είναι τα πράγματα. Και πιστεύω πραγματικά ότι η Ευρώπη δεν μπορεί βεβαίως να γνωρίσει αυτή την πραγματικότητα και πρέπει να έχει τη δική της θέση. Όταν μιλάμε για τη στρατηγική αυτονομία, αυτό συνδέεται με αυτό που είπαν και πολλοί από εσά, ε, ότι εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό ε, σε ό,τι αφορά το, ε, τα φάρμακα, το φαρμακευτικό υλικό, πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από ό,τι πιστεύαμε και σε κρίσιμες περιστάσεις όπως αυτή αυτό φαίνεται και πρέπει βεβαίω να ενισχύσουμε αυτήν τη στρατηγική αυτονομία να μπορέσουμε ταυτόχρονα να προσπίσουμε τις αξίες μας, ε, τα συμφέροντά μας όσο γίνεται πιο αυτόνομα. Αυτό δεν σημαίνει, όπως είπα, ίσες αποστάσεις, το είπα νωρίτερα. Ε, πρέπει να είναι σαφές όμως το τι θέλουμε, το τι περασπιζόμαστε, το είτε μας αρέσει είτε όχι. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε πάντα με τις ΗΠΑ, ε, διότι οι ΗΠΑ παίρνουν μονομερείς αποφάσεις με τις οποίες εμείς δεν συμφωνούμε. Εφόσον λοιπόν δεν συμφωνούμε, δεν μπορούμε να τους υποστηρίξουμε οι αποφάσει που παίρνουν παραδείγματο χάρη για το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο ε, και φαντάζομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί εδώ. Πρέπει ταυτόχρονα να διατηρήσουμε την διατλαντική αυτή σχέση ε, και διότι συμμεριζόμαστε και το ίδιο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό ε, λέμε ότι έχουμε συστημική αντίθεση με την Κίνα, διότι δεν έχουμε το ίδιο πολιτικό σύστημα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ε, σε όλα και πάντα να είμαστε απέναντι στην Κίνα. Ε, διότι υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα όπου χρειάζεται συνεργασία. Στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. Ε, κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι κεντρικές απαντήσεις. Ναι, για τα όπλα υπόθηκε νωρίτερα κάτι. Προφανώς και εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει έτσι μια κούρσα εξοπλιστική, αλλά ε, απ' την άλλη υπάρχουν ε, σειράξεις ε, που πρέπει να αντιμετωπιστούν και εκεί δυστυχώς χρειάζονται και όπλα. Την επόμενη φορά που μια ομάδα τρομοκρατών θα επιτεθεί σε ένα χωριό στο Μάλι και θα εκτελέσουν όλους τους κατοίκους θα τους στείλουμε ένα κείμενο ψηφίσματος για να τους πούμε να μην συνεχίσουν να το κάνουν. Ε, εγώ νομίζω ότι είναι πιο λογικό οι δυνάμεις αυτών των χωρών και οι δικέ μα, τη βοήθεια των δικών μα δυνάμεων για την αντιμετώπιση τη τρομοκρατία να έχουν τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Τελείωσε έτσι εδώ πέρα η συζήτησή μας ε, για αυτό το θέμα. Θα ακολουθήσουν οι ψηφοφορίες για τον θέμα του Χονγκ Κόνγκ και για την ανάγκη να υπερασπιστούμε την αυτονομία του Χονγκ Κόνγκ αύριο. Οπότε κλείνει εδώ η κοινή συζήτηση και συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη σε λίγο. Can we start? Yes. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζεται η συζήτηση. Πριν γίνει αυτό, ξεκινάει ο πρώτος γύρος ψηφοφοριών από τις 10.30 μέχρι τις 11.45. Θα έχουμε την ίδια διαδικασία όπως και χτες όλες οι ψηφοφορίες θα είναι ονομαστικές. Μπορείτε να δείτε στο, ε, έγγραφο, στο έγγραφο τα ψηφοδέλτια. Οι δηλώσεις ε, μπορούν να γίνουν γραπτός. Θα γίνουν δεκτές όμως δηλώσεις με ένα όριο 400 λέξεων. Άρχεται η ψηφοφορία, μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι τις 11 και 45. Τα αποτελέσματα αυτής της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 2 και 4. Οπότε, τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Έχουμε δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής πολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με την COVID-19 και αντίκτυπο στην ελευθερία της έκφρασης. Να υπενθυμίσω ότι δεν θα γίνουν δεκτές μπλε κάρτες και η διαδικασία του ΚΕΤΘΙΑ και ξεκινάμε με την εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την κυρία Μπρίζετς. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ε, η κρίση αυτή η υγειονομική που αντιμετωπίζει ο κόσμος ε, έχει επιδεινωθεί από άλλη μια επιδημία. Οι πολίτες μας αντιμετωπίζουν λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες που δημιουργούν σύγχυση αλλά και διακινδυνεύουν τις ζωές και την υγεία τους. Το Συμβούλιο λοιπόν έχει τονίσει την ανάγκη να εντείνουμε τις προσπαθίες μας κατά της παραπληροφόρησης, να υπάρξει μια στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και των κοινωνικών πλατφορμών. Υπάρχει μια συνένεση στο Συμβούλιο για την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση χωρίς να εμποδίζουμε την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα, η συντονισμένη δράση μας ε, πρέπει να συντονίζεται με τις δημοκρατικές αξίες μας, την ελευθερία έκφρασης και τα ελεύθερα μέσα όλα τα κράτη-μέλη, τα θεσμικά τους όργανα και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την επιδημία αυτή. Πάρα πολλά έχουν γίνει στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Η Task Force Στρατηγικής Επικοινωνίας που είχε φτιάχτη πριν τις ευρωεκλογές παρακολουθεί την παραπληροφόρηση. Η συνολική προσέγγιση απαιτείται σε όλα τα επίπεδα για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της παραπληροφόρησης. Αυτό σημαίνει παρακολούθηση και ανάλυση της παραπληροφόρησης, ε, της χειραγώγησης, επιβολή των κανόνων προστασίας δεδομένων, προσπάθειες να ενισχύσουμε τα πλουραλιστικά μημιέ, ενημέρωση για τα μημιέ και των πολιτών. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις πλατφόρμες για να επιτευχθούν υψηλότερες ε, προδιαγραφές διαφάνειας και λογοδοσίας για να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Επίσης, ε, θα πρέπει ακριβώ να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με το να εκθέτουμε τα πραγματικά γεγονότα. η Προεδρία παίρνει πάρα πολύ στα σοβαρά την παραπληροφόρηση σε σχέση με τον κορονοϊό και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε συνενή συνεργασία κρατών μελών, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και φορέων και διεθνών οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Από τις 28 Ιανουαρίου ενεργοποιήσαμε το κέντρο πολιτικής αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπου συνευρίσκονται διάφοροι εμπειρογνώμονες ε, των κρατών μελών ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα πολιτικής προστασίας και δημόσιας υγείας. Είδαμε εκεί και το ζήτημα της παραπληροφόρησης και θεωρούμε ότι οι αυτές θα μπορούσαν να διαταράξουν την χαλάρωση του εγκλισμού και την προσπάθεια για να ανακαλυφθεί ένα εμβόλιο. Δίναμε τις προσπάθειές μας και στην οριζόντια ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσουν οι χώρες τις υβριδικές απειλές στην Πολιτική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ασφαλείας. Είχαμε επίσης βίντεο διασκέψεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας. Υποθέτουμε ότι η παραπληροφόρηση θα συνεχίσει να υφίσταται, θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα εσωτερικά και εξωτερικά. Η παραπληροφόρηση αυτή επιδεινώνει τις υφιστάμενες ε, διαφορές ε, στην Ανατολική Γειτονία και στα Δυτικά Βαλκάνια. Στην ε, σχετική σύνοδο κορυφή 26 Μαΐου, οι ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Δυτικών Βαλκανίων συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα τη παραπληροφόρηση και άλλων τέτοιων δραστηριοτήτων. Όπω είπα, στην αρχή. Όταν πολεμάμε την παραπληροφόρηση δεν πρέπει να ξεχνάμε την ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος των πολιτών να ενημερωθούν και να διασφαλίσουμε την ελευθερία λόγου και των μημιών. Μετά την πανδημία αυτή, πάρα πολλά κράτη-μέλη ενέκριναν ευρύτατα μέτρα που στόχο είχαν να μπορέσουν να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών τους. Πολλά από αυτά τα μέτρα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα, δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να δυσφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν αναλογικά προ τον σκοπό με χρονικό περιορισμό και θα μπορούν να υφίστανται δημοκρατικό έλεγχο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για λογοκρισία ή για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει οι κυβερνήσεις να στηρίξουν τα ανεξάρτητα ΜΜΕ που είναι σύμμαχοί μας στην καταπολέμηση του κορονοϊού. Η δημοκρατική συζήτηση, η ελευθερία των ΜΜΕ και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή. Η προστασία αυτών των αξιών είναι προτεραιότητα για το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Υφυπουργέ. Έχουμε σήμερα την μεγάλη τιμή να έχουμε δύο αντιπροέδρους της ε, Κομισιόν για την συζήτηση αυτή. Τον είπα το εκπρόσωπο τον κύριο Μπορέλ ε, και την ε, αντιπρόεδρο την κυρία Γιούροβα. Χαιρόμαστε πολύ. ποιο. θα ξεκινήσει ο κύριος Μπορέλ. Έχετε τον λόγο. Thank you, Madam Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Είναι προφανές ότι η πανδημία, ο ιός ε, της πανδημίας συνοδεύτηκε και από μια πανδημία παραπληροφόρησης. Είχαμε πολλές πληροφορίες παραπλανητικές και αυξήθηκαν οι δραστηριότητες ξένων παραγόντων με στόχο την παραπληροφόρηση. Τι μπορούμε να κάνουμε. Η παραπληροφόρηση μπορεί να δημιουργήσει τεράστια ζημιά όσον αφορά την πανδημία που έχει να κάνει με την υγεία. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι ακόμα πιο επικίνδυνο. Είχαμε παραπληροφόρηση που έλεγε ότι πίνοντα χλωρίνη, για παράδειγμα, ε, αντιμετωπίζει τον ιό. Και εδώ δεν, δεν, δεν θέλω να πω Δεν εννοώ τίποτα άλλο εκτό από αυτό που λέω. Πιείτε χλωρίνη και είσαστε ασφαλεί. Ή ότι δεν βοηθάει το πλήσιμο των χεριών. οδηγεί όμως και στο έγκλημα. Ε, βανδαλισμοί σε βάρος ε, εξουπλισμού 5G. Θυμόσαστε τι έγινε. Το Μάρτιο του 2020 οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν από την Επιτροπή και τον είπα το εκπρόσωπο να αναλάβει δράση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ανακοίνωση για την παραπληροφόρηση σε σχέση με την πανδημία και με τη συνάδελφο και αντιπρόεδρο επίσης συμπληρώσαμε την ανακοίνωση αυτή, η οποία συνοψίζει βασικά το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα για να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση όσον αφορά την πανδημία. Οι πληροφορίες προφανώς και ενημέρωση δεν έχουν σύνορα. Ξέρουμε ποιοι ήταν οι στόχοι. Οπότε επιτρέψτε μου τώρα να στραφώ στην εξωτερική διάσταση η πανδημία έτυχε εκμετάλλευση από διάφορους φορείς, κρατικούς και μη κρατικούς. Από τη Ρωσία, για παράδειγμα, που κυκλοφόρησαν διάφορες πληροφορίες ε, συνωμοσία με στόχο την Ευρωπαϊκή Ένωση και γείτονε χώρες όσον αφορά την έλλειψη αλληλεγγύης και γενικά δημιουργήθηκε σύγχυση. Και η Κίνα συμμετείχε. Η Κίνα μπορεί να είναι κάτι καινούριο, η Ρωσία ήταν πιο δραστήρια, αλλά κινέζικες πηγές πρόθεσαν την εικόνα αυτή που τους παρουσίαζε σαν το πιο τέλειο σύστημα, που πιο τέλεια αντιμετώπισαν την πανδημία με το δικό τους το σύστημα για να αντιμετωπίσουν την κρίση κορονοϊού. Ε, φυσικά υπάρχει μια παραπαγάνδα, ο καθένας μπορεί να θέλει να λέει ότι τα κάνει καλύτερα από τους άλλους, αλλά άλλο πράγμα είναι να λες ότι πιστεύεις ότι είσαι ο καλύτερος και άλλο είναι να τα βάζεις όμως με τους άλλους και να προσπαθείς να τους διχάσεις. Υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνος από κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν την πανδημία σαν άλοθη για να περιορίσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή την ελευθερία έκφραση. Στην προηγούμενη συζήτηση κάποιοι από εσά αναφερθήκατε σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά και πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Τι έχουμε κάνει για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι τάσει. Προωθούμε την επικοινωνία και τη στρατηγική στα Δυτικά Βαλκάνια, στην γειτονιά μας ε, γενικά. Προσπαθήσαμε από πλευρά τη Επιτροπή να το κάνουμε, δημοσιεύσαμε εκθέσει. Ενημερώσαμε για τις τάσεις αυτές, μοιραστήκαμε τα ευρήματά μας με άλλους εταίρους μας, με χώρες, την κοινωνία των πολιτών κτλ. Όσοι εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν επιτελέσουν ένα πολύ δύσκολο και ιστορική σημασία έργο επ' αυτού. Χρησιμοποίησαμε καλά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση αυτή με τα συστήματά μας, τα οποία συνδέουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με τις χώρες μέλη αποδείχτηκε ένα δίκτυο αυτό πολύτιμο. Και έχουμε δημιουργήσει ειδικό χώρο για την ανταλλαγή πληροφορών όσον αφορά την παραπληροφόρηση αυτή σε σχέση με τον ε, κορονοϊό. Επίσης έχουμε ενισχυμένη συνεργασία με τους διεθνείς μας ε, τέρους και χρησιμοποιούμε το μηχανισμό ε, γρήγορης ανταπόκρισης και επίσης ενισχύσαμε και τις σχέσεις μας με τον ΟΙΕ. Τώρα στο μέλλον θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις δράσεις μας αυτές με στρατηγική επικοινωνία και ανακοινώσεις, με ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές και ενεργο, ενεργοποιώντας πιο γρήγορα τα συστήματά μας τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση. Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, με τον ιδιωτικό τομέα, ε, παρατηρώντας τι γίνεται με τις παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών κλπ. Έχουμε το πρόγραμμα για τη σταθεροποίηση της ειρήνης που περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση ε, κρίσεων σε περιοχές που είναι πιο ευάλωτες. Δεν χρειάζεται να μπω περισσότερο σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να μιλήσει η Αντιπρόεδρος για την ε, διαφάνεια, η κυρία Βέρα Γιούροβα, η οποία θα σας παρουσιάσει ε, το έργο που γίνεται στις κοινωνικές πλατφόρμες και άλλες πτυχές του ζητήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Τον λόγο έχει η κυρία Γιούροβα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, μόλις ακούσαμε από τον Τζοζέπ Μπορέλ τις βασικές παράμετρους ε, για αυτό που ονομάζουμε infodemic, ε, μια πανδημία παραπληροφόρησης δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν ε, αποφασίσαμε ε, να προετοιμάσουμε μια ανακοίνωση με τίτλο «Τα σωστά δεδομένα, τα ακριβή δεδομένα». Διότι είναι σημαντικό να ενημερώσουμε για το τι συνέβη ως τώρα ε, απέναντι στις πληροφορίες αυτές, διότι στα πλαίσια του COVID δεν ξεκινήσαμε από το μηδέν να πολεμούμε την παραπληροφόρηση. Είχαμε ήδη κάποιες βέλτιστες πρακτικές, είχαμε το σχέδιο δράσης και βεβαίως θελήσαμε επίσης ε, να ε, προετοιμάσουμε ένα κατάλογο για το τι πρέπει να κάνει ο καθένας ε, και αναφέρομαι σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων και οι πλατφόρμες και οι πληροφορίες μας έχουν να κάνουν με τρία στοιχεία. Οι πηγές παραπληροφόρησης, ποιοι τις διωγγώνουν και τις μεταδίδουν και ποιοι είναι οι στόχοι. Ο Ζωζέπ προηγουμένω αναφέρθηκε στις ξένες πηγές παραπληροφόρησης και χαίρομαι που το ανέφερε αυτό διότι πιστεύω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση της Γεωπολιτικής μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο αν είμαστε στεναροί. Πρέπει όμως και εμείς στο εσωτερικό μας να κοιτάξουμε τα του οίκου μας, τα της επικοινωνίας μας. Πρέπει και η δική μας ιστορία ε, για την Ευρώπη και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού να περάσει. Και ήρθε η ώρα ε, να το κάνουμε εμείς αυτό, να μην αφήσουμε άλλους να ε, καλύψουν το χώρο αυτό. Σε ό,τι τώρα τους διάβλους επικοινωνίας και παραπληροφόρησης, ιδιαίτερα οι πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Καλωσορίζω τα μέτρα που έχουν πάρει αυτές οι πλατφόρμες στα πλαίσια της κρίσης και τη δέσμευσή τους. Είναι απαραίτητη αυτή η δέσμευση. Το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε στις πλατφόρμες αυτές και από κοινού έχουμε αυτόν τον κώδικα καλών πρακτικών βοήθησε έτσι ώστε να έχουμε πιο γρήγορα αυτές τις νέες πολιτικές. Συμφωνήσαμε στις πλατφόρμες ότι θα προωθήσουν links προς την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, προς τις αρχές υγείας γενικότερα και θα αποσύρουν όσα ε, όσα παραπληροφερούν ή αυξάνουν ε, τις τιμές προϊόντων ή κάποια επικίνδυνα πράγματα που έχουν ε, υποθεί και αναφέρθει ο Ζωζέπ. Αυτό έφερε αποτέλεσμα. Η Google, παραδείγματος χάρη, ε, μπλόκαρε ή απέσυρε πάνω από 18 εκατομμύρια διαφημίσεις που σχετίζονται με το κορονοϊό. Βεβαίως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ε, και αυτός ο κώδικας είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε διαφάνεια και λογοδοσία. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πώς φτάνουν οι πληροφορίες σε αυτούς και από πού προέρχονται η κοινή μας ανακοίνωση ζητεί από τις πλατφόρμες να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους και μηνιαία να μας ενημερώνουν για τις δράσεις τους έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα παραπληροφόρησης που σχετίζονται με το COVID-19. Όχι προς την Κομισιόν, προς το κοινό, προς το ευρύ κοινό, έτσι ώστε να μπορούν να ξέρουν όλοι τι συμβαίνει στο διαδίκτυο. Οι στόχοι τώρα. Ε, Βεβαίω εμείς είμαστε οι στόχοι αλλά και οι πολίτες, οι πολίτες της Ευρώπης. Ε, το να λέει κανεί ψέματα δεν είναι κάτι καινούριο ούτε φοβίζει από μόνο του. Αυτό που με φοβίζει είναι να όταν, όταν, πιστεύουμε εύκολα τέτοια ψέματα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο προσεκτικοί ε, ως κοινωνία, να υποστηρίζουμε τα, ελεύθερα μίντια, τα ανεξάρτητα μίντια, τα μίντια τα οποία ελέγχουν τα δεδομένα. Ε, σύντομα θα έχουμε και ένα σχέδιο εκπαίδευσης ε, ε, για τα ζητήματα αυτά και θα υπάρχει ένα κεφάλαιο για το πώ θα είμαστε πιο ανθεκτικοί, πώ θα έχουμε μια πιο κριτική σκέψη σε ό,τι αφορά την πληροφορία που λαμβάνουμε. Εμεί θα υποστηρίξουμε ε, τι ε, δραστηριότητε έρευνα και ελέγχου των δεδομένων μέσω του σχετικού παρατηρητηρίου για τα μίντια. Ε, αργότερα αυτό το μήνα θα δοθούν 9 εκατομμύρια ευρώ για τα σχετικά hub στα κράτη-μέλη, θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε και για την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του λόγου. Είναι πολύ βασική αρχή. Όταν υπάρχουν ε, νομοθεσίες για ποινές, ε, για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και αυτές οι νομοθεσίες είναι πολύ ασαφείς και καλύπτουν υπερβολικά πολλά πράγματα, τότε ε, αυτό δυσκολεύει το έργο των δημοσιογράφων. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Δημιουργεί, ε, ε όπως αντιλαμβάνεστε, έλλειψη δημοκρατίας και έλλειψη ελευθερίας. Ε, είναι κάτι που οδηγεί ε, σε μια λάθος προσέγγιση. Χρειαζόμαστε ανοιχτά, ελεύθερα μίντια, σωστή ενημέρωση και ανθεκτικές δημοκρατικούς, δημοκρατικούς θεσμούς στους οποίους μπορεί να εμπιστεύονται. Ιδάλλως οδηγούμαστε σε λογοκρισία. Ε, δεν θέλω να δημιουργήσω ένα Υπουργείο, Υγείας, ε, Υπουργείο Αλήθειας. Συγγνώμη. Ξέρετε ότι ζούσα σε ένα σύστημα πριν από το 1989 όπου υπήρχε μόνο μία επίσημη αλήθεια, δεν υπήρχε πλουραλισμός ε, στα μίντια, δεν υπήρχε ελευθερία σκέψης ή λόγου. Ε, χρειαζόμαστε μια ανταγωνιστική, πλουραλισμος στα μιλια αγορά σκεψης η λογου Είναι απαραίτητο αυτό στη δημοκρατία ε, Στι δημοκρατίε, όπω και στον τομέα του καταγωνισμού γενικότερα, όπου οι καταναλωτέ ε, επιφελούνται από αυτή την ελεύθερη ανταγωνισμό, έτσι και οι πολίτε επιφελούνται από την ελεύθερη, ε, τον ελεύθερο ανταγωνισμό του ελεύθερου λόγου. Είναι το πρώτο σκέλος της απάντησής μας στην παραπληροφόρηση αυτή η προσπάθεια. Υπάρχει και η νομοθεσία για τι ψηφιακέ υπηρεσίε, υπάρχει το σχέδιο δράση για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, όπου θα μιλήσουμε για το παράνομο και το επιβλαβέ υλικό στο διαδίκτυο που οδηγεί στην παραπληροφόρηση και πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα ε, το γεγονός ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ε, να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή που έχετε δημιουργήσει εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι η συνεργασία αυτή ε, θα είναι, ελπίζω, επικοδομητική για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Περνάμε τώρα στη συζήτηση με τον πρώτο γύρο των κοινοβουλευτικών ομάδων. Ξεκινάει ο κύριος Μπίλτσικ για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπετεκπρόσωπε, κυρία Υπουργέ. Η κατάσταση με το COVID-19 έχει τονίσει ότι η παραπληροφόρηση σκοτώνει ανθρώπους αλλά και την δημοκρατία. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την διάδοση ψευδών ειδήσεων πολύ πιο συστηματικά. Καλωσορίζω τα σχέδια για να ενταθούν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, αλλά χρειάζεται πιο έντονη προσπάθεια για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης από Ρωσία και Κίνα. Πρέπει να μιλήσουμε με μια ενιαία ενωμένη ευρωπαϊκή φωνή κατά της Ρωσίας και της Κίνας που θέλουν να υπονομεύσουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Αλλά η μάχη κατά της παραπληροφόρησης δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής. Χρειάζεται έντονη δράση ε, κατά των πλατφορμών που διαδίδουν την παραπληροφόρηση. Καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν για να δίνουν αναφορά κάθε μήνα οι πλατφόρμες για το τι κάνουν. Χρειάζεται λοιπόν σαφής και νομοθετική δράση που θα διασφαλίσει ότι όλες οι πλατφόρμες θα φέρονται υπεύθυνα και θα αναφέρουν το τι κάνουν για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση. Για το καλό της ασφάλειας των πολιτών μας ε, θα πρέπει να διακρίνουμε τα γεγονότα από τα ψέματα, την επιστήμη από τα ψέματα και τους δημοσιογράφους από τους σκιτζίδες. Ε, αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπίλτσιτς. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η κυρία Πύρη έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η διάδοση τη ε, παραπληροφόρηση και των ψευδών ειδήσεων είναι απειλή κατά τη δημοκρατία μας, υπονομεύει τι δημοκρατίε μα, βλάπτει τι αξίες μα και τα συμφέροντά μας. Αλλά κατά τη διάρκεια μιας πανδημία, όπως είπε ο υπουργό, ε, κινδυνεύουν πλέον ζωέ, Αλλά ούτε αυτό δεν έχει σταματήσει τις ξένες δυνάμεις από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ο αριθμός των εκστρατιών αυτών από την Ρωσία και την Κίνα ήταν τεράστιος οι παρεμβάσει και ο υβριδικό πολεμό δεν πρέπει ποτέ να είναι στρατηγική, αλλά ειδικά κατά τη διάρκεια μια παγκόσμια υγειονομική κρίση. Η ανακοίνωση τη Κομισιόν είναι άλλο ένα σημαντικό βήμα προ μια συνολική στρατηγική κατά των ξένων παρεμβάσεων. Χρειαζόμαστε αυστηρότερε ρυθμίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στόχο διαφόρων δράσεων και πρέπει ανάλογη να είναι και αντιδρασή μα. Οι σοσιαλδημοκράτες είναι στο προσκήνιο του αγώνα αυτού. Θα προτείνουμε λοιπόν την σύσταση μια επιτροπή κατά των ξένων παρεμβάσεων και τη παραπληροφόρηση. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο για να προστατεύσουμε τι δημοκρατίε μα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να παίξει αυτόν τον ρόλο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ακολουθεί ε, η κυρία Πάρνσαντούα για το Ρινιό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πότε υπήρξε πιο πολύ παραπληροφόρηση συμβαίνει όταν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή το κοινοβούλιο δεν είχαν αντιδράσει ακόμα αποτελεσματικά και συνολικά και όχι αρκετά αποτελεσματικά στην πανδημία. Αυτό ήταν το ευάλωτο σημείο μα και από αυτό υποφελήθηκαν όσοι προχώρησαν σε παραπληροφόρηση. Γιατί υπάρχει μια στρατηγική αποδυνάμωσης του κράτου δικαίου, των δημοκρατικών μα συστήματα ε, συστημάτων. Και όταν έχουμε ένα δύναμο σημείο με χίλιο πτέρνα, ακριβώ εκεί πάνε και χτυπάνε όσοι θέλουν να προχωρήσουν σε παραπληροφόρηση. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι φανατισμένοι, είναι θυσμένοι στο ψέμα. Σαν ε, νέοι στρατιώτες σε ένα νέο πεδίο μάχης που είναι το διαδίκτυο. Και αυτές οι ομάδες χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο και αποδυναμώνουν την ιδεολογία και τις δημοκρατίες μας. Και αυτό είναι το σοβαρό. Συνεπώς, φωνάζουν πιο πολύ, τρομοκρατούν και εμείς πρέπει να στηρίξουμε την ελευθερία έκφρασης, έναν καθαρό χώρο και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία του φανατισμού. Αυτή που λειτουργούν σαν στρατιώτες της παραπληροφόρησης δεν ξέρουν το κακό που κάνουν, ενώ αυτοί που το θέλουν και το καθοδηγούν βεβαίως και το ξέρουν και μας κάνουν μεγάλο κακό. Γι' αυτό πρέπει και να το αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Ντεμάν για το ομάδα ID. Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε έναν επικίνδυνο δρόμο. Όλο και περισσότερα κράτη απειλούν τα θεμέλια της δυτικής δημοκρατίας, δηλαδή την ελευθερία γνώμης. Και όταν οι Ευρωπαίοι Επιτροπή μιλάνε για Action Plan Against Information, μια task force, ένα σύστημα συναγερμού και ε, προειδοποιούν ε, τον ε, ιδιωτικό τομέα για την παραπληροφόρηση. Βεβαίως θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα ελέγχουν την ακρίβεια των ειδήσεων. Λοιπόν, και Όλα αυτά βεβαίως γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τα χέρια των παραδοσιακών κομμάτων και μιμιέ και το καθιστός ανησυχεί. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω να σταματήσετε με αυτήν την υφέρπουσα λογοκρισία. Ζήτω οι διαφορετικές απόψεις. Ζήτωσαν. Σας ευχαριστώ Λαγκοντίνσκι για την ομάδα των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πρέπει να είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξει ποτέ μια μαγική λύση για το θέμα της ε, παραπληροφόρησης, αλλά τέλος πάντων στην πολιτική είμαστε και γνωρίζουμε πως ε, δεν υπάρχει μαγική λύση για τα πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς όσον αφορά την αφετηρία. Η αφετηρία είναι να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, όχι να την βλάψουμε. Γι' αυτό η στρατηγική μας θα πρέπει να είναι τριπλή και συνολική. Πρώτα απ' όλα να πολεμήσουμε τις γεωπολιτικές επιθέσεις από το εξωτερικό δεύτερο να ενημερώσουμε τους καταναλωτές τύπου και διαδικτύου και τρίτον, να προστατεύσουμε την προσωπική άποψη και τον ελεύθερο λόγο. Βλέπουμε τις παγίδες που αντιμετωπίζουμε. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βεβαίως ε, απέδειξαν μια στιβαρή στάση και σωστά τα είπε ο κύριος Μπέικρουλ. Είναι και μια μάχη διαφορετικών αφηγημάτων. Απ' την άλλη μπορούμε να πέσουμε σε μια αντιδημοκρατική παγίδα. Γι' αυτό η ποινικοποίηση της παραπληροφόρησης όπως έγινε στην Ουγγαρία ή στην ε, Πολωνία. Η δίωξη εκπροσώπων φαρμακευτικών εταιριών στη Βουλγαρία επειδή ήθελαν να προειδοποιήσουν ε, για την έλλειψη φαρμάκων. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα δεν πρέπει να ξεχνάμε τις στρατηγικές μας αρχές. Αντιμετωπίζοντας ε, την παραπληροφόρηση πρέπει να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, όχι να την καταστρέψουμε και κάτι άλλο, γιατί ε, πάρα πολύ το ξεχνάνε. Η ανωνυμία στο διαδίκτυο είναι θετικό. Προστατεύει τις γυναίκες, τις μειονότητες, τους αντιπολιτευόμενους. Γι' αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να καταργηθεί. Κάτι ακόμα για την εκπαίδευση. Πρέπει να επενδύουμε περισσότερο στην εκπαίδευση στα ζητήματα δικαιοσύνης ε, και αξιών και να μην τα περικόψουμε κατά 20% και θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινωνία των πολιτών και να μην την αγνοούμε. Έτσι θα προστατεύσουμε τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Μπουσαντεβιλιάλμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ζει μια κρίση αξιοπιστία μετά τη νίκη του Brexit του 2016. Κάποια κράτη-μέλη, κάποιοι θεσμοί τη Ένωση έχουν. Θεωρούν ότι η έλλειψη αξιοπιστία έχουν να κάνουν με παραπληροφόρηση από εξωτερικού ή εσωτερικού παράγοντε. Ξεχνούν, ξεχνούν όμω ότι η παραπληροφόρηση δεν προέρχεται μόνο από εκεί, ούτε είναι κάτι καινούριο. Τα ψέματα πάντα υπήρχαν και συνήθω προέρχεται από την εξουσία. Προέρχεται από την εξουσία. Ξέρετε ότι στην πρώτη σελίδα ε, του, της, του, της βίβλου μαθαίνουμε πως ε, το φίδι ξεγελάει τον Αδάμ και την Εύα. Μιλάμε για παραπληροφόρηση όμως ή μιλάμε για λογοκρισία και να τελειώσουμε τελικά με την ελευθερία έκφρασης. Δεν πρέπει αυτές οι υπηρεσίες που ε, ελέγχουν τα δεδομένα να μα λένε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα και να λαμβάνουν κρατικέ ενισχύσει γι' αυτό, διότι είναι ιδιωτικέ εταιρείε που έχουν τα δικά του οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Η κρίση του κορονοϊού μα έδειξε ότι κανεί δεν είναι αλάθητο. και εκεί υπήρξε παραπληροφόρηση από όλου. από την Κίνα, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία, τι ίδιε τι κυβερνήσεις και τα μίντια. Το να πιστεύει κανεί ότι στο κοινοβούλιο αυτό θα πρόκειται εμεί να φτιάξουμε την αλήθεια, να την κατασκευάσουμε, είναι, είναι ασυγχώρητο. Είναι ασυγχώρητο ατόπιμα ε, και υπεροψία. Θα συνεχίσαμε με τον κύριο Λαγό, αλλά δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Οπότε περνάμε στον κύριο Τόμακ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι Καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα, πέρα από την κρίση του κορονοϊού, είχαμε να εντοπίσουμε και ένα άλλο σοκ. Την πανδημία σε επίπεδο παραπληροφόρησης. Είναι πραγματικό σοκ, διότι δεν μπορούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να κρύβουμε την αλήθεια. Τα fake news προέρχονται από τη Ρωσία. Εμείς που ζούμε στη Ρουμανία, στην Πολωνία, στις χώρες της Βαλτικής, ξέρουμε πόσο ειδικεύεται η Ρωσία στην παραπληροφόρηση. Και αυτή η επίθεση, κύριε Μπορέλ, είναι μια πολύ σκληρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Και αυτό που είπατε είναι σωστό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια, μια δέσμευση. Πρέπει όμως και να απαντήσουμε